διάταξη αυτό το θέμα. Οπότε έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη αυτή τη εβδομάδα. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξη, έκθεση της κυρίας Λάρα Κόμη για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Η κυρία Κόμη λοιπόν έχει τον λόγο, η συγκεκριά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Προέδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτέλους φτάσαμε στην τελική συζήτηση και την οριστική έγκριση αυτού του σημαντικού κανονισμού. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι προσωπικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη δουλειά που έγινε και τη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και όλους τους και όλους εκείνους που μίλησαν και παρενέβησαν και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πλευράς ε, Συμβουλίου. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιπλέον φτάσαμε και στην έγκριση ενός χαρτοφυλακίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορική αγορά εντός ενός έτους και έχουμε και μία έγκριση και συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση έτσι επιταχύνοντας την όλη νομοθετική διαδικασία. Μπορώ να πω πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι πρόκειται επί πραγματικής ε, επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέβαλε τα μάλα στον καθορισμό του τελικού κειμένου του κανονισμού. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου ε, ενισχύεται σίγουρα και εύχομαι αυτό το σημαντικό θεσμικό όργανο και εκείνοι που εκπροσωπούνται, δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες, να μπορούν στο μέλλον να έχουν όλο και περισσότερη εμπλοκή και συμμετοχή. Τώρα θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές ιδιαίτερες του κανονισμού και να υπογραμμίσω τη σημασία που έχουν οι αλλαγές που έγιναν. Πάνω απ' όλα, με τη θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού. Μια στιγμή κύριε και κύριοι, δεν μπορεί κανείς να ακούσει την εισηγήτρια. Εάν δεν θέλετε να μιλήσετε στη συζήτηση αυτή, παρακαλώ να εγκαταλείψετε ήσυχα την αίθουσα. Μια στιγμή, κυρία Κομή. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα υπογραμμίσω συντομία κάποιε ιδιαιτερότητε του κανονισμού για να διαφανούν οι σημασίες, η σημασία που έχουν οι αλλαγέ. Ε, τη θέση σε ισχύ πάνω από όλα αυτού του κανονισμού το σύστημα θα εξακολουθεί να εδράζεται επί αρχών παγιωμένων, δηλαδή εθελοντικό το σύστημα ε, στο ιδιωτικό τομέα και θα βασίζεται επί της ε, αρχής της κόρης εξουσίας στα κράτη-μέλη. Δεν θέλαμε να χαλάσουμε ένα σύστημα που λειτουργεί και λειτουργήσε αρκετά καλά. Θέλαμε όμως να εντοπίσουμε τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να γίνει πιο δημοκρατικό το σύστημα και πιο ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα. Εξασφαλίσαμε εξάλλου και την πιο ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή των stakeholders ε, των φορέων συμφερόντων που έχουν και σημασία το δημόσιο τομέα και στη φάση της διαβούλευσης πριν από την επεξεργασία της εντολής και ακολούθως. Πρόκειται επί σημαντικότητα του σημείου διότι αυτό αυξάζει το δημοκρατικό χαρακτήρα του συστήματος και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των προτύπων όλοι οι ενδιαφερόμενοι και από την αγορά, εκπρόσωποι και τον δημόσιο τομέα. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η διαβούλευση να γίνεται σε όλες τις φάσεις τη διαδικασία. Και γι' αυτό το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινοποίηση που επιτρέπει στους stakeholders να καταχωρηθούν και μετά αυτομάτως να ενημερώνονται. Είναι σωστό να εξασφαλίζεται η συμμετοχή στο σύστημα αυτό των επιχειρήσεων και των εκπροσώπων των δημοσίων συμφερόντων. Εξίσου σημαντικό όμως να εξασφαλίζεται και η παρουσία στη διαδικασία των αρχών και των δημοσίων αρχών ε, στο διοικητικό τομέα και στο νομοθετικό τομέα. Και κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η απλούστευση του τρόπου συμμετοχής των. Εγώ ήθελα πολύ να το πετύχω αυτό εντός του κανονισμού κυρίως σε εθνικό επίπεδο, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λόγω της μειωμένης διάστασή τους και λόγω των γλωσσικών προβλημάτων έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στο σύστημα, αλλά αποτελούν όμω την πραγματικότητα την οικονομική βάση του ευρωπαϊκού μα συστήματο. Το ευρωπαϊκό επίπεδο μετά πρέπει να συμβάλλει στην εξασφάλιση αυτή τη εκπροσώπηση που εν πρώτη θα πρέπει να ξεκινά από κάτω. Δηλαδή να ακολουθούμε το σύστημα από κάτω προ τα άνω. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων τη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση με το διεθνές επίπεδο που είναι από τους μεγάλους στόχους ε, που έχουμε θέσει. Διότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει και να δώσει τα πρότυπά τη σε παγκόσμια κλίμακα και έτσι να γίνουν αυτά παγκόσμια πρότυπα. Ξεκίνησε ένα σημαντικό ε, διάλογο με τι Ηνωμένε Πολιτείε με την ε, αποστολή που έγινε στη Ουάσιγκτον που πήγε εκεί η Επιτροπή ΙΜΚΟ και θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως αρνήθηκε το αίτημα του Συμβουλίου να υπάρξουν ε, εφαρμοστικές ε, πράξεις όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τις τεχνολογίες για την επικοινωνία και την πληροφόρηση. Ε, διότι θεώρησαν ότι θα ε, επιβραδινόταν η όλη διαδικασία γιατί θα ήταν μεγάλο ο φόρτο εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω το Κοινοβούλιο εξασφάλισε μια φάση διαβούλευση πριν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αν χρειάζεται να καθοριστούν τεχνικές προδιαγραφέ. Λοιπόν, φτάνω στα συμπεράσματα και μπορώ να πω ότι ο κανονισμό απλουστεύει το όλο σύστημα από πλευρά διοικητική και οικονομική εξασφαλίζοντα υψηλότερο επίπεδο διαφάνεια. Παραδείγματο χάρη, μα αγάγει τη δημοσίευση ιστοσελίδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή του καταλόγου των προτύπων των εναρμονισμένων, που αποτέλεσαν αντικείμενο μια απόφαση επίσημης. Ε, δεν θα μακρηγορήσω, διότι και άλλες... είναι πάρα πολλές σημαντικές πτυχέ και δεν θέλω να μπω στις τεχνικέ λεπτομέρειε. Και ήταν πάρα πολύ περίπλοκο το όλο θέμα. Δηλαδή, αφήνω λοιπόν χώρο για τη συζήτηση και είμαι στη διάθεση όλων για δίποτε διευκρίνηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Κόμη. Η Επίτροπος, η κυρία Ρέντινγκ, έχει τώρα το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο αμέλη, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Λάρα Κόμη, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, για την εσωτερική αγορά και την προστασία του καταναλωτή και ειδικότερα τον πρόεδρό της, τον κύριο Μάλκομ Χάρμπουρ, για την πολύ σημαντική δουλειά που έχουν κάνει. Η τυποποίηση είναι ένα από τα βασικά εργαλεία ε, που στηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομία. Η συνεργασία μεταξύ των χρηστών, ε, της, της βιομηχανίας, αλλά και των δημοσίων αρχών, αλλά και των υπηρεσιών τυποποίησης, όλη αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική ε, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τελικά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας οδήγησε στην εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι έτσι ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ενισχύεται και η διαλειτουργικότητά τους, κάτι το πολύ σημαντικό για να είναι ανταγωνιστικές και να μπορέσουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα και ε, υπηρεσίες. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα πρότυπα είναι βασικό εργαλείο ώστε να προσελκύσουν και να ε, διατηρήσουν τους καταναλωτές ως πελάτες τους. Και φαίνεται ότι οι καταναλωτέ ικανοποιούνται όλο και περισσότερο από την χρήση ενιαίων προτύπων. Το ίδιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει διότι έτσι επιτυχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Πέρα από όλα αυτά, όλη αυτή η τυποποίηση και ενοποίηση των προτύπων πρέπει να ανταποκριθεί στι καινούργιε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε μπροστά μα. Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, στη σύγκληση των τεχνολογιών, ε, στην προστασία του καταναλωτή, στη βελτίωση τη προσβασιμότητα, στην ε, ε, βελτίωση τη προσβασιμότητα κυρίω για άτομα με αναπηρίε. Τον Ιούνιο του 2011 υιοθετήθηκε αυτό το πρώτο πακέτο μέτρων και χαίρομαι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή συζητά για την υιοθέτηση του κανονισμού ε, για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Είναι το τελευταίο κομμάτι αυτού του πακέτου και με αυτό το κανονισμό θα λυθούν τρία βασικά προβλήματα. Πρώτον, το γεγονός ότι ζητήθηκε να χαραχθούν πρότυπα ε, είναι πολύ σημαντικό και έτσι η νομοθεσία θα βελτιωθεί μέσω του ετησίου προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω της οικονομικής στήριξης που προσφέρεται. Δεύτερον, θα συμπεριληφθεί ε, η ευρωπαϊκή τυποποίηση παντού η γνώμη των φορέων της αγοράς δεν ακούγεται πολύ μέχρι σήμερα. Με τον κανονισμό αυτό θα έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των φορέων των κοινωνικών φορέων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και κατά τρίτο λόγο ε, θα βελτιωθεί η κατάσταση με τις ε, δημόσιες αγορές και τις συμβάσεις. Ξέρετε, ε, πολύ συχνά παγκόσμια φόρουμ είναι αυτά τα οποία κάνουν αντίστοιχες ανακοινώσεις και όχι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την τυποποίηση και έτσι οι προδιαγραφές που επιβάλλονται δεν ταιριάζουν με τη δική μας κατηγορία προτύπων τα οποία λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τις κρατικές αρχές όταν αυτές προκυρήσουν διαγωνισμούς. Επομένως τώρα θα έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης και έτσι οι αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις νέες προδιαγραφές υπό τον όρο ότι θα πληρούνται συγκεκριμένα ε, κριτήρια που συνάδουν με τις αρχές τυποποίησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Βάσει του κανονισμού θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο πολιτικής την ε, ε, τυποποίηση και την ενοποίηση των προτύπων και στον τομέα των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και πολλοί στο Κοινοβούλιο, λυπάται για την αιμονή του Συμβουλίου να επιβάλλει ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες επιτροπολογίας, οι οποίες, ε, των οποίων η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθεί σε αυτή την περίπτωση και οι οποίες είναι και αρκετά χρονοβόρες. Γι' αυτό το λόγο θα αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη ρήτρα αναθεώρηση την οποία ευτυχώς έβαλε το Κοινοβούλιο σε αυτό το κείμενο ώστε να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε νέες προτάσεις μέσα σε δύο χρόνια. Ωστόσο, δεδομένου του γεγονότος ότι τα βασικά στοιχεία της αρχικής πρότασης έχουν γίνει δεκτά και ε, προσπαθώντας να λειτουργήσουμε επικοδομητικά, να επιτύχουμε συμβιβασμό, να υπάρξει ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή θα δεχθεί το κείμενο έτσι όπως προτείνεται μεταξύ Συμβουλίου ε, και Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνάδελφε Γκέρεκ, για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι απαιτήσει αυτές για τυποποίηση είναι κάτι σημαντικό για την οικονομία κλίμακας, για την ποιότητα και για την ασφάλεια των καταναλωτών. Η τεχνολογική πρόοδος είναι ταχύτερη από τη θέσπιση προδιαγραφών και προτύπων και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να καθορίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά τα πρότυπα. Αυτό θα διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς. Θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Άρα θα πρέπει να έρθουν υπάρχοντες φραγμοί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί εναρμόνιση. Τυποποίηση πρέπει να εμπλέκει και τους οργανισμούς εθνικούς τυποποίησης. Αλλά αγνοούνται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης. Χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας και των διάφορων εθνικών οργανισμών. Ευχαριστώ. Τώρα εν ονόματι των πολιτικών ομάδων στους αγορητές, ξεκινώντας με τον συνάδελφο ΣΒΑΠ για τέσσερα λεπτά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση για την Ευρωπαϊκή τυποποίηση έχει συζητηθεί ήδη αρκετά και θεωρώ πως παρόλες τις δικαιολογημένες αντιρρήσεις της Αντιπροέδρου της κυρίας Ρέντινγκ μπορούμε να πούμε εδώ πέρα πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα αυτά τα οποία σχετίζονται με την ομοθεσία εσωτερική αγορά του κυρίου Μπαρνιέ έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μπορώ να σας πω λοιπόν αγαπητοί συναλφοί, το γιατί εγώ θα συγχαρώ την κυρία Κομή. Πρώτα απ' όλα κατάφερε αυτό το οποίο ζητούσαμε στο παρελθόν συχνά, δηλαδή να ε, γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, δηλαδή τους κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν άμεσα στο εθνικό δίκαιο και όχι οδηγίες. Δεύτερον, κατάφερε να ενισχύσει τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί στο παρελθόν μόνο το Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο μπορούσε να σταματήσει ε, προτάσεις τυποποίησης. Ενώ με αυτό το οποίο συζητάμε τώρα και θα ψηφίσουμε αύριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να σταματήσει προτάσεις τυποποίησης εάν παραδείγματος χάρη Υπάρχουν παραδείγματο χάρη προτάσει τυποποίηση για κάποια κτίσματα τα οποία είναι παράνομα όπω ε, υπήρχαν σε ορισμένα κράτη-μέλη. Κατόπιν ε, Βεβαίω διαπιστώνουμε πως θα πρέπει να παραμένουν οι κανονισμοί προσανατολισμένοι προς την αγορά, να έχουμε βεβαίω μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, οι οποίοι όμως δεν θα καθορίζουν τις στις προδιαγραφές αυτές και βέβαια θα υπάρξει και ένα σύστημα ειδοποίησης τρίτων γιατί βεβαίως θα πρέπει αυτά και να τα παρατηρεί η κοινωνία, να τα αποδέχεται η κοινωνία, να τα ελέγχει η κοινωνία και μπορούμε εδώ πέρα να εγγυηθούμε με αυτή την πρόταση πως και οι αρχές ε, και όλοι όσοι συμμετέχουν θα έχουν πλήρη πρόσβαση εδώ πέρα και κάτι το οποίο είναι σημαντικό και αφορά όλες τις ομάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλήρη πρόσβαση όσον αφορά την ρύθμιση του ε, δικού τους ε, των κανόνων που τους αφορούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως ε, αυτό είναι μόνο ένα μόνο μέτρο από τα 12 μέτρα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν για μια πλήρη εσωτερική αγορά, οπότε δεν πρόκειται για ένα ορόσημο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απλά ένα κομμάτι και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία να προχωρήσουμε και στην ε, πράξη της ενιαίας αγοράς υπαριθμών 2 και θεωρώ πως θα συμφωνήσει εδώ πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Συνάδελφε Σάλτεμος, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Øh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ μίλησα, για... μίλησα στους εκλογείς μου για το θέμα αυτό της υποποίησης και δύσκολα μπορούσαν να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Αλλά βεβαίως μπορούμε να πούμε πως η υποποίηση και το έργο αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία για την ευρωπαϊκή συνεργασία γιατί βεβαίως χωρίς την τυποποίηση θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Παραδείγματο χάρη τι γίνεται. Δεν θα ξέραμε ποιο στικάκι USB είναι συμβατόν ποιον υπολογιστή και τα λοιπά. Και τις λάμπες ε, πυρακτώσεως και τις μπρίζες ε, και τα λοιπά. Τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Αφορούν προδιαγραφές λοιπόν για όλα τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Και βεβαίως το θέμα αφορά και τα τρόφιμά μας και το περιβάλλον το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε και είναι σημαντικό λοιπόν να αναθεωρήσουμε την ομοσία που υπάρχει, να επανεξετάσουμε τις προδιαγραφές που υφίστανται να υπάρξει και μια απλοποίηση και για τις επιχειρήσεις και για την εσωτερική αγορά. Αυτά είναι τρία πράγματα τα οποία είναι σωστά σε αυτή την πρόταση και τα οποία βρίσκω θετικά. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερη διαφάνεια στην ε, νομοθετική αυτή διαδικασία και να δούμε και ποια εντολή υπάρχει προς αυτό. Αλλά είναι επίσης αποφασιστική σημασία στο να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή στο έργο αυτό. Και αυτό ήταν αποφασιστική σημασία για εμάς σοσιαλιστές και δημοκράτες. Για να συμπεριλάβουμε δηλαδή και ΜΚΟ για να μπορέσουν όλοι να πούν την γνώμη τους για τα θέματα της τυποποίησης, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε πώς θα εργαζόμαστε άνοιχτά, πώς ε, θα εφαρμόσουμε την εντολή την οποία έχουμε. Μιλάμε και για τις αρμόδιότητες των κρατών μελών, αλλά κυρίως μιλάμε για τις γενικές αρχές, την κοινωνική ασφάλιση, όλα αυτά τα οποία πρέπει να τηρηθούν και βεβαίως ε, Νομίζω πως οι δικές μας ε, τροπολογίες οδήγησαν στο ότι διαφυλάσσονται και οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, οπότε έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αμοιβαία επωφελής και έχουν ε, πάρα πολύ μεγαλύτερο ρόλο τώρα οι διάφορες οργανώσεις. Είναι τα πράγματα λοιπόν απλούστερα, γρηγορότερα και πραγματικά θέλω να συγχαρώ και τους ε, καταναλωτές ε, και τις επιχειρήσεις ε, αλλά και τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω σε εσά το λόγο, συνάδελφε Μάντερ. Α, δεν βλέπω να είναι στη θέση του συνάδελφο. Συνάδελφε Ρούλε, για τρία λεπτά για την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη, θα επικεντρωθώ στα βασικά. Οι προδιαγραφές είναι κάτι το σημαντικό, είναι ένα μέσο, κωδικοποιούν σε μια τεχνική βάση, σε μια τεχνική γλώσσα την ε, η ευρωπαϊκή αγορά και προωθούν έτσι την καινοτομία. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση έχει αποδεικτεί επιτυχημένη και σε καιρού οικονομική κρίση θα πρέπει να εξυγχρονίζουμε προσεκτικά τα μέσα αυτά χωρί να διακινδυνεύει η ουσία του. Νομίζω τα καταφέραμε αυτό. Έχουμε επίσης διασφαλίσει την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σημαντικών κοινωνικών ομάδων και άρα βελτιώσει και την αποδοχή τους αλλά βεβαίως χωρίς την εθελοντική αυτή συνεργασία ε, πρέπει να δούμε χωρίς την οποία θα υπήρχε διαδικασία πρέπει να δούμε ποιος θα επομιστεί το κόστος της ε, συμμετοχής θεωρώ λοιπόν πως θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει πιο πολύ σε αυτόν τον τομέα αλλά αποδέχομαι το συμβασμό ο οποίος επιτεύχθηκε Επίσης, η τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών επεκτάθηκε ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες της βιομηχανίας ε, και στον τομέα της πληροφορικής. Ταυτόχρονα βεβαίως ήταν σημαντικό στον τομέα των υπηρεσιών να μην περιορίσουμε τα ελεύθερα επαγγελματά και το δημιουργικό δυναμικό που υπάρχει εκεί πέρα. Παραδείγματο χάρη η τυποποίηση είναι ένα παράγοντα κόστους και άρα θα πρέπει να υπάρχει μόνο εκεί όπου έχει σημασία για την αγορά και θεωρούμε πως μια πλατφόρμα με συμμετέχοντες όλους του ενδιαφερόμενους θα φροντίσει για την κατάλληλη διαβολή. Τέλο για εμάς ήταν ε, ο διαχωρισμό μεταξύ τυποποίηση και νομοθεσία. Δεν θέλουμε νομοθεσία από την πίσω πόρτα ως κοινοβούλιο. Σε γενικέ γραμμές νομίζω λοιπόν πως είχαμε έναν καλό συνδεσμό και αύριο θα τον υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ECR. Συνάδελφοι Κόζουσνη και έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω το εξής. Αυτή η συζήτηση για το πακέτο αυτό των μέτρων τυποποίησης πράγματι είναι μια μεγάλη επιτυχία και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από αυτή την έννοια συγχαίρω την εισηγήτρια διότι κατάφερε ε, να φέρει σε πέρα στη δουλειά της με πολύ ε, καλό τρόπο. Μπράβο Λάρα λοιπόν για όλα αυτά. Η τυποποίηση είναι πράγματι στοιχείο κλειδί ώστε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση των προτύπων και να ενισχύσουμε την αντιγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Θα πρέπει να δούμε και τις ε, νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα ICT. Νομίζω ότι πράγματι θα είναι εργαλείο αυτό για να στηρίξουμε όλο αυτό το κλάδο, τον ICT. Η τυποποίηση είναι για να έχουν, είναι πολύ σημαντική για να έχουν όλη πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Και μπορούμε και να βασιστούμε στην οδηγία για τις υπηρεσίες άλλωστε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Πάσκα, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερως την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει το ε, περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να ε, ε, ενημερώσουμε, να βελτιώσουμε τις αρχές για την τυποποίηση. Καλό θα είναι να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των αλλαγών όμως δεν γίνεται αναφορά στις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης. Δηλαδή δεν γίνεται αναφορά στην αρχή της εθνικής εκπροσώπησης. Δεν γίνεται αναφορά σε αρχές ε, που αναφέρονται στην αναστολή και στην πάυση των διαδικασιών. Και γενικά πολλά άρθρα έχουν μια πολύ γενική διατύπωση και επιδέχονται πολλών και διαφορετικών ερμηνεών. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες της Επιτροπής Έρευνας και Βιομηχανίας αλλά και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Οι άλλοι αγορητές έχουν το λόγο. Συνάδελφε Μπάστος, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω Συγχαίροντα την κυρία Κόμη, την εισηγήτρια, έξοχη δουλειά τη είναι πάρα πολύ σημαντική, ζωτική σημασία για το μέλλον τη Ευρώπη. Σε έναν κόσμο και σε μια κοινωνία που επιταχύνονται οι αλλαγέ, χρειαζόμαστε πραγματικά ένα σύστημα για να συμπεριλαμβάνει επίκαιρε τυποποίησει, επίκαιρε προδιαγραφέ και θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, να βελτιώσουμε τη ζωή των καταναλωτών με αυτόν τον τρόπο και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική ένταξη, μεγαλύτερη τεχνολογική προόδος, διασύνδεση μεταξύ δικτύων και συστημάτων, κυρίως σε τομείς όπου αναμειγνύεται η τεχνολογία της πληροφορικής. Όπως αναφέρθηκε, χρειάζεται μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι κρισίμου σημασίας για να είναι πιο σύγχρονη η ενιαία αγορά και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε για τη θέσπιση προδιαγραφών, ούτως ώστε να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα και να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό που συζητούμε τώρα ακολουθεί αυτές τις γραμμές. Η συγγήτρια προσπίζεται αυτούς τους στόχους και σωστά. Ε, αποφεύγει τον κατακαιρματισμό που δημιουργεί αύξηση κόστου συναλλαγών, μεγάλες δαπάνες ενισχύει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία τυποποίησης, κυρίως στο εθνικό επίπεδο, και διευκολύνει την πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στις προδιαγραφές, ενισχύεται η συμμετοχή ε, των εκπροσώπων κοινωνικών συμφερόντων, τους καταναλωτές, τους περιβαλλοντολόγους, τους εργαζομένους ανθρώπους, οι άνθρωποι με αναπηρίες μπορούν όλοι αυτοί να συμμετέχουν στη θέση των προδιαγραφών. Εκπροσωπούν το κοινό, το δημόσιο συμφέρον. Αυτή η έκθεση θα συμβάλλει στην επαναπρόθεση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Καινοτομία, για την ενίσχυση τη Ευρώπη και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μα. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε Γκέπχαρτ, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι για να αναφερθώ και εγώ στο παράδειγμα της κυρίας Σάλντε Μόζα, ας υποθέσουμε πως υπάρχει ένα USB και ο κάθε υπολογιστής έχει διαφορετική πρόσβαση και σύνδεση και ο καθένας χρειάζεται ανταπτοράκι. Μόνο αυτό το παράδειγμα σας δείχνει πόσο σημαντική είναι η τυποποίηση στην καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων τις οποίες διευκολύνει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα μας αυτό. Επίσης καταφέραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιφέρουμε πάρα πολλές βελτιώσεις στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια όσο και την ε, σκιώδη εισηγήτρια οι οποίες έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε δύο θέματα παρά το ότι ο χρόνος πιέζει τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς. Πρώτον έχουμε τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς και να φροντίσουμε ώστε η τυποποίηση και οι προδιαγραφές να μην γίνονται μόνο από τους μεγάλους αλλά να λαμβάνουν υπόψη και τα συμφέροντα των μικρών γιατί ο κίνδυνος είναι σε αυτές τις περιπτώσεις οι μεγάλοι να επιβληθούν και οι μικροί να χρειαστεί να ακολουθήσουν κάτι το οποίο κοστίζει και καταφέραμε λοιπόν να υπάρξει στήριξη και χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα. Το δεύτερο θέμα που ήταν σημαντικό για εμάς ήταν η εξαίρεση ενός μέρους των υπηρεσιών που ε, εντάχθηκαν πλέον στον τομέα της τυποποίησης. Μιλάμε για τις υπηρεσίες που έχουν γενικό οικονομικό ενδιαφέρον και βεβαίως εδώ πέρα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα ελεύθερα επαγγέλματα γιατί η τυποποίηση μπορεί να είναι ακόμα και επικίνδυνη γιατί μιλάμε για ευελιξία, για δημιουργικότητα που θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και νομίζω πως καταλήξαμε σε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό και μπορούμε να συμφωνήσουμε ως ομάδα αλλά όπως σας είπα έπρεπε να γίνει πολλή δουλειά και νομίζω στο μέλλον να ελπίζω στο μέλλον να είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Γκάλ Πέλτς, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια. Να συγχαρώ και την ε, εισηγήτρια η οποία νομίζω έφερε επιτυχώς εις πέρας το έργο της. Όσον αφορά την τυποποίηση, συμφωνώ, πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία, αλλά πρέπει να πω πως η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται να αποβεί εις βάρος της ποιότητας. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να επιταχυνθεί το διοικητικό σκέλος αυτής της ε, διαδικασίας, οι αρχές τυποποίησης ε, πρέπει να το κάνουν αυτό από κοινού με κάποιον συμβασμό και βέβαια να υπάρχει και διαφάνεια. Θεωρώ πως η Κομισιόν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματο χάρη με την επιτάχυνση της ε, διαδικασία αρχής και τέλους, με την υπογραφή των συμβάσεων, με την πιστοποίηση των υπηρεσιών. Συμφωνώ επίσης με αυτό το οποίο είπε η εισηγήτρια, θα πρέπει δηλαδή να βασιστούμε στις υφιστάμενες δομές και θεωρώ πως η <clears throat> πρόσβαση στην ε, πιστοποίηση δεν αφορά μόνο την τιμή των ε, πρωτογραφών αλλά και οι εθνικές αρχές τυποποίησης θα πρέπει εδώ πέρα να συμπεριληφθούν έτσι θα μειώσουμε το κόστος και θα καταλήξουμε ε, σε ένα πακέτο τυποποίησης με μικρότερη τιμή βεβαίως. Σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν εδώ πέρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λοιποί συμμετέχοντες. Εγώ θα έλεγα πως δεν υπήρχαν ε, και καμιά φορά εμπόδια, απλά δεν ενδιαφέρονταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ήταν το κόστος ε, αυτό το οποίο τις εμπόδιζε και ήταν κάπως παθητικές. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό, να βρούμε τις μεθόδους για να κινητοποιήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εμπλακούν εδώ πέρα. Γιατί αυτό συνεισφέρει και στην ε, ανταγωνιστικότητα και στην αηφορία της Ευρώπης. Και ε, νομίζω πως μπορούμε όλοι να στηρίξουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Βάιλερ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ναι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάπου τα γελιά μου εδώ πέρα βλέχτηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδης εισηγητές για το έγγραφο αυτό το οποίο θα εγκρίνουμε αύριο. Αναφέρθηκαν πάρα πολλά πράγματα για τη χρησιμότητα της ε, τυποποίησης. Να αναφέρω και εγώ δύο ε, παραδείγματα. Την, ε, τον φορτιστή για τα κινητά, τον ενιαίο δηλαδή φορτιστή για τα κινητά και τη, τα ηλεκτρικά οχήματα. Χωρίς τυποποίηση δεν θα γινόταν τίποτα. Βεβαίως δεν είναι γνωστό το πώς βγαίνουν οι προδιαγραφές. Δεν το κάνει το Κοινοβούλιο, ούτε στο μέλλον θα το κάνει, αλλά εθνικές και ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές και Ινστιτούτα όπως η ΣΕΝ και η ΣΕΝΕΛΕΚ τα κάνουν αυτά. Τα τελευταία 25 χρόνια ήταν βεβαίως μια καλή εποχή, αλλά υπάρχει και μια σειρά ελλημάτων και ελλείψεων. Ήταν η διαδικασία αργή, ακριβή, αδιαφανής, χωρίς συμμετοχή. Με την πρόταση αυτή νομίζω το αλλάξαμε αυτό και θα γίνει και πιο φτηνή η πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έχουμε τα συνδικάτα, τις οργανώσεις των καταναλωτών, την σύνδεση με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και χαίρομαι βεβαίως και για την εμπλοκή του τομέα των δημοσίων προμηθειών. Τέλος, για την αποδοχή από την κοινή γνώμη. Πρέπει να δούμε τι ε, γίνεται, γιατί ξέρετε πως το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης, το γνωστό DIN, ε, είχε μεγάλες επιφυλάξεις. Ε, για παραδείγματος χάρη στο κρατήδιο της ΕΣΥΣ, ε, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν επίσης επιφυλάξεις, αλλά νομίζω πως με αυτή την πρόταση είναι όλοι ικανοποιημένοι. Νομίζω λοιπόν πως θα τα καταφέρουμε και στο μέλλον να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στους αγορητές ε, που ζήτησαν την προσέγγιση της προσοχής Προέδρου, Catch Μάτζι Κουκόβιτς, συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στη διαδικασία της αναβάθμισης του συστήματος τυποποίησης. Ξέρω τι σημαίνει τυποποίηση τι σημαίνει η διαδικασία αυτή για μια επιχείρηση. Πολύ δύσκολη ήταν. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν συμβάλλει στη βελτίωση για την κατάσταση των επιχειρήσεων. Και όσον αφορά τα ICT, ας έχουμε υπόψη ε, τον Bill Gates ε, που είχε πει εδώ και 10 χρόνια ότι με κάθε λύση για να βρει κάποια, όταν βρίσκει κάποια λύση σκέφτεται πρώτα πώς θα την τυποποιήσει. Και έτσι η Microsoft δημιούργησε λύσεις και προέβαινε στην αναβάθμιση. Να πω και κάτι για τις υπηρεσίες. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία με Ινδία, Ρωσία και άλλες αναπτυσσόμενες αγορές στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Τσικάου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ η ευρωπαϊκή τυποποίηση πράγματι κάνει πιο ανταγωνιστικό τον κόσμο των επιχειρήσεων όταν ανταποκρίνεται στο παγκόσμιο σύστημα η τυποποίηση. Τα πρότυπα, οι κανόνε, είναι πολύ σημαντικό για να είναι ανταγωνιστικέ οι επιχειρήσει και κυρίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η συμμετοχή του λοιπόν στη διαδικασία διαμόρφωση των προτύπων είναι απαραίτητη. Οι κανόνε και τα πρότυπα θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να προσφέρουν καινοτόμε λύσει σε όλη αυτή αυτή την προσπάθεια και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική συμμετοχή θα είναι αποτελεσματική εάν μειωθεί το κόστος και αρθούν οι γλωσσικοί φραγμοί. Καλό ε, θα είναι να γίνει προσπάθεια να δοθεί ενδεχομένως και δικαίωμα ψήφου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν συμμετέχουν στους οργανισμούς τυποποίησης. Η Επιτροπή Ήτρε έχει εξετάσει διάφορα συστήματα ε, καθορισμού των ε, τελών και των ε, τιμών με μειωμένες τιμές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις βιοτεχνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Κομφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να στραφώ, εν συντομία, προς την κυρία Επίτροπο. Είπατε, και συμφωνώ, ότι το έργο της ηγήτριας ήταν ε, έξοχο. Πιστεύω ότι και οι επιτροπές συνέβαλαν να εμπλουτίσουν επικαιροποιώντας αρχική πρόταση. Υπάρχουν καινοτόμα στοιχεία σίγουρα στο τελικό κείμενο, όπως η συμμετοχή των stakeholders στη διαδικασία λήψης απόφασης, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις προδιαγραφές, η εισαγωγή της κοινωνικής ρήτρα. Ε, ε, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγνώριση της πλατφόρμας των multi-stakeholders Όλες αυτές είναι συνιστώσει που δίνουν αξία και ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Όμως πιστεύω ότι όσον αφορά τις υπηρεσίες, το σημείο ισορροπία που εξευρέθη πρέπει να εκτιμηθεί, πρέπει να εγκριθεί, αλλά χρειάζεται όμως στο μέλλον ε, να έχουμε μια νέα ρύθμιση που να επιτρέπει διαδικασία εναρμόνισης χωρίς αυτό να επιβαρύνει τους πολίτες ή να γίνει ένα στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών συστημάτων. Λοιπόν, η δουλειά που έγινε είναι πολύ καλή, με πολύ συνέπεια, αλλά ήδη από τώρα ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η διαδοχική φάση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Χάρμπορ έχει το λόγο. Uh, uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, θέλω πως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής, να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής που εργάστηκαν τόσο σκληρά για αυτό το θετικό αποτέλεσμα που είναι πραγματικά βελτίωση για ένα σημαντικό κομμάτι της ενιαίας αγοράς. Και πρέπει να θυμηθούμε απόψε και οπωσδήποτε θα ε, το ήθελε και η κυρία Επίτροπος πως πρόκειται για την πρώτη από τις δεσμεύσεις για την ε, πράξη της ενιαίας αγοράς αυτή η οποία περνάει και θα ψηφιστεί αύριο. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω πως δεδομένης της σημασίας του θέματος και του μεγάλου ενδιαφέροντος ε, από χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπλέκονται στη διαδικασία τυποποίησης, πώς λάβαμε μία απόφαση όλοι οι συντονιστές ε, να κάνουμε βεβαίως ε, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό ως παρασκευαστικό έργο δηλαδή μια στρατηγική έκθεση για τις προδιαγραφές πριν από 18 μήνες και μας έδωσε τη δυνατότητα να διαβουλευτούμε πριν περάσουμε στην νομοθεσία. Νομίζω πως συνεισέφερε αυτό στην ποιότητα της δουλειάς και είναι κάτι το οποίο γνωρίζω πως ε, το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι από άλλες επιτροπές, είναι εδώ πέρα συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Εμπορίου και βεβαίως αυτό δείχνει την σημασία που αποδίδουν στο θέμα αυτό της τυποποίησης. Γι' αυτό είμαι σίγουρος πως αύριο βεβαίως θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η έκθεση, αλλά αντικατοπτρίζει νομίζω τη σημασία του θέματος στο ότι εναπλάξαν εδώ πέρα τόσες πολλές ομάδες πολιτικές. Ε, Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Μάντερς, θέλετε να μιλήσετε έτσι όλος εξαιρετικά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και με συγχωρείτε για την καθυστέρηση έμπλεξα στην κίνηση. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την κίνηση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Λαρακόμη για την συνεργασία και βεβαίω αυτά τα οποία είπε ο κύριο Χάρμπορ είναι εξαιρετική η συνεργασία και θεωρώ πως είναι καλό το αποτέλεσμα που έχουμε για τη βιομηχανία, για την οικονομία, για τον καταναλωτή και πως εμείς ως Ευρώπη Νομίζω πως έτσι θα μπορούμε ευκολότερα να θέσουμε τις παγκόσμιες προδιαγραφές και θα μετράει ως οικονομική ήπειρος η Ευρώπη στον ε, κόσμο. Και αυτό θα γίνει ευκολότερα με την τυποποίηση. Βεβαίως ε, είναι ε, κάτι το εθελοντικό και βεβαίως μην ξεχνάμε πως πριν από χρόνια είχα συζητήσει τότε με τον κύριο Φερχόιγγεν ε, την πρόταση για τους φορτιστές για τα ε, κινητά τηλέφωνα και για τις υπόλοιπες φορητές συσκευέ τα iPads παραδείγματος χάρη κάτι το οποίο βεβαίως θα κάνει πάρα πολύ ευκολότερη τη δουλειά για τη βιομηχανία και για τον καταναλωτή. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για τον κόπο τον οποίο κάναμε. Σας ευχαριστώ. Η Επίτροπος, η κυρία Ρέντινγκ, έχει το λόγο. Euh, Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα μου ε, θέσατε, το τελευταίο μάλιστα από τον κύριο Μάντερς. Να πω ότι υπάρχει εθελούσια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιομηχανίας για την εναρμόνιση των ε, τελών ε, και των τιμών. Και αυτό όντως είναι πολύ σημαντικό και θα ε, ωφελήσει ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Ως προς το πρώτο ερώτημα για την τυποποίηση των υπηρεσιών, να πω στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο κανονισμός επιβεβαιώνει ε, τη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αξιοποιήσει την τυποποίηση των υπηρεσιών ως εργαλείο πολιτικής για την εναρμόνιση μεταξύ των διαφορετικών κλάδων. Τούτων λεχθέντων. Συμφωνώ απολύτως με τα λόγια ε, του Προέδρου κ. Μάλκομ Χάρμπορ. Πράγματι, είναι το πρώτο από τα 12 ενδεχομένως βήματα που πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη που θα έχει ο καταναλωτής ε, και να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία έχουν υιοθετηθεί στο κείμενο της Επιτροπής του 2011. Είναι καλό για τη βιομηχανία, για τους καταναλωτές, για την οικονομία. Ωστόσο, ε, κάτι το οποίο έχουν επισημάνει πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελούν όλα αυτά εξέλιξη και όχι επανάσταση. Ο κανονισμός ε, ε, η οικοδομή πάνω στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να έχουμε ένα ενιαίο διαφανές περιεκτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολιτικές εδώ στην Ευρώπη αλλά και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, θέλω λοιπόν ε, να καλέσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζικά να ψηφίσουν υπέρ ε, στη ψηφοφορία για αυτό το, το πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Δίνω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια. Λάρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη συζήτηση μέσω της οποίας παρουσιάσαμε έναν κανονισμό με έναν τρόπο πλήρη. Διεφάνισαν τα πιο σημαντικά σημεία. Αυτός ο κανονισμός θα εγγυηθεί στις εθνικές αγορές και στην ευρωπαϊκή αγορά καλύτερη διάδραση, εξασφάλιση μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, κάτι που χρειάζεται η Ευρώπη, βελτίωση όλου του συστήματο ε, της διαμόρφωσης των προτύπων, διευκολύνει και κάνει αποτελεσματικότερη τη δουλειά των επιχειρήσεών μα. Αυτές οι προδιαγραφές έχουν συνέπειε για του πολίτες. Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφο. Σελντεμόζε. Ε, βελτιώνουν τη ζωή τους. Θα πρέπει να το κάνουμε κατανοητό αυτό και στους συναδέλφους μας για να μπορέσουμε να διαδώσουμε και στην εντός Ευρώπης αυτή την άποψη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα θα είναι ανταγωνιστικό σε ε, ε, εθνικό επίπεδο. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ανδρέα Σβάμπ ότι χρειάζονται περισσότεροι κανονισμοί και λιγότερες οδηγίες αν θέλουμε έχουμε πραγματικά μια εσωτερική αγορά όπως πρότεινε ο Καθηγητή Μόντι και όπως πρότεινε και ε, ο Επίτροπος Μπαρνιέ, διότι αυτή είναι η σωστή οδός για να πετύχουμε μια ένωση που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά που είναι μια ένωση πολιτική και στο τέλος μπορούμε να την αποκαλέσουμε και ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ, κυρία Κόμη. Πέρα τη συζητήσεως, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τώρα στην ημερήσια διάταξή μας έχουμε την έκθεση ακούνια που αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηδών. Δίνω παρευθύ το λόγο για ένα τετράλεπτο στην εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό